Buenos días. Καλημέρα σας. Αν συμφωνείτε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Ladies and gentlemen, please. Quiet. Try to start. Buenos días. Vamos a... Καλημέρα σας. να ξεκινήσουμε ένα πρωινό με πολλές ψηφοφορίες. Πριν να περάσω όμως την έγκριση την ημερήσια διάταξη, επειδή έχουμε πάρα πολλές ψηφοφορίες, να προσπαθήσουμε να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί για να μην χρονοτριβούμε, σας παρακαλώ. Λοιπόν, για να ολοκληρώσουμε την ψηφοφορία γρήγορα, εγώ δεν θα λέω τόσε ψήφοι υπέρ, τόσε ε, κατά κτλ. Θα βλέπετε τα αποτελέσματα στι οθόνε. Εγώ απλώ ε, θα αναφέρομαι στον αριθμό τη Τροπολογία, θα λέω αν εγκρίνεται ή αν απορρίπτεται. Και αν υπάρχει κάποια αμφιβολία θα ζητάτε το λόγο. Αλλά νομίζω θα είναι πιο εύκολο να το κάνουμε έτσι και τα αποτελέσματα θα τα βλέπετε στην οθόνη. Έτσι λοιπόν μπορούμε να κινηθούμε πιο γρήγορα. de votación. Έχετε όλοι τις κάρτες για να ψηφίσετε. <laughs> να σας ε, ομολογήσω όλοι, όλοι μάλλον έχετε τις κάρτες εκτός από τον πρόεδρο. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την έγκριση της ημέρης της διάταξης. Υπάρχουν κάποιες αλλαγές, θα σας τις γνωστοποιήσω. Για το σημείο 10, την έκθεση Το σημείο 11, Καντέκ. 17, Πατράου και στις 14 θα αναβληθούν για την επόμενη συνεδρία της Επιτροπής. Το 10, 11, 17 και 14. Δεν θα τα συζητήσουμε τα σημεία αυτά σήμερα. Συμφωνείτε? Και επίσης να σας υπενθυμίσω ότι από τις 5 το απόγευμα και μετά θα έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων με την Επιτρόπο Δαμανάκη θα είναι και κλεισμένων των θυρών. Και επί της αρχής θα μας ενημερώσει η κυρία Επίτροπος για τις συμφωνίες με τρίτες χώρες και για τις ανεξέλιξη διαπραγματεύσεις. Προέρχεται αυτό σε συνέπεια με μια συνεδρίαση που είχαμε με την κυρία Επίτροπο όπου γνωστοποιήθηκε η γενική δυσαρέσκεια της κομισιό της Επιτροπής Και συνήθως έρχονταν ο κύριος Ντεπίπερ και κάναμε εδώ αυτή τη συνεδρίαση και κλείμανε των θυρών. Όμως ε, εγώ δήλωσα τη δυσαρέσκεια της Επιτροπής μας ότι δεν μαθαίναμε και πάρα πολλά σε αυτές τις συνεδριάσεις, δεν απαντούσα οι αρμόδιοι της Επιτροπής σε καμία από τις ερωτήσεις που έθετε η Επιτροπή μας. Έτσι λοιπόν έπρεπε ή να εγκαταλείψουμε αυτές τις συνεδριάσεις ή να τις κάνουμε δημόσια. Έτσι λοιπόν αποφάσισε η κυρία Δαμανάκη να παρευρεθεί εδώ, να μας εξηγήσει πώς πάνε οι διαπραγματεύσεις και να απαντήσει σε όλα. Αυτή είναι λοιπόν, αυτός είναι ο σκοπός της σημερινής συνεδρίασης το απόγευμα. Κατόπιν έχουμε την έγκριση των πρακτικών τη 21 η Μαου 2012. Αν δεν υπάρχει αντίρρηση, εγκρίνουμε τα πρακτικά. Περνάμε στο σημείο 3, ανακοινώσει του Προέδρου. Δεν έχω κάποια συγκεκριμένη ανακοίνωση, πέρα από αυτά που σας είπα. Και, αν συμφωνείτε, να περάσουμε στο σημείο 4, κοινή οργάνωση αγορών στον τομέα προϊόντων αλίας και υδατοκαλλιέργειας. Ο κύριο Στίβενσον είναι ο εισηγητή και να ξεκινήσουμε με τις ψηφοφορίε έτσι όπως σας είπα. Και θα διευκρινίσω και τη δική μου ψήφο. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Μπορούμε να ξεκινήσουμε. Τροπολογία 72. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. να επαναλάβουμε. Είστε όλοι έτοιμοι. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε. Πέρας. Se rechaza la propuesta. Ah, ça commence mal. Bueno, comenzamos. Vamos a ver. Λοιπόν, για να δούμε. Έχετε όλοι βάλει σωστά τις κάρτες. Λοιπόν, επαναλάβουμε την ψηφοφορία, να ξεκινήσουμε. Αλλά αφού δείτε ότι λειτουργούν οι κάρτες, μην τις ξαναπειράξετε, γιατί αν ένα λεπτό χρειαζόμαστε για κάθε ψηφοφορία τροπολογίας, αύριο θα τελειώσουμε. Λοιπόν, τροπολογία 72, άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε. Σε <laughs> Πέρας. Απορρίπτεται. Λοιπόν, δεν ψηφίζουμε την 73, 75. Έρχεται ψηφορία. Πέρας. Απροβάδα. Εγκρίνεται. 76. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 77. Άρχεται η ψηφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Η NV7 είναι ταυτόσιμη. Περνάμε στην 78. Άρχεται η ψηφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 82. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Επαναλαμβάνουμε. Λοιπόν, αν πάω γρήγορα να μου το πείτε. Περνάμε στην 82. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. 24 hanno votato, a Silofese non lo so. Hay una más. Aquí 24 han votado, 25 Hay un, hay un voto más de los socialistas. Sí. Grupo socialista. Έχει, υπάρχει μία ψήφος παραπάνω από τους σοσιαλιστές. Να επαναλάβουμε την ψηφοφορία για την 82, τροπολογία 82. Αλλά να προσπαθήσουμε στο μέτρο του δυνατού να μην ε, τροποποιούμε τις ομάδες και όσους ψηφίζουν. Διαφορετικά θα είναι αδύνατο. Λοιπόν, για να δούμε. Για τελευταία φορά. Τροπολογία 82. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Συνεχίζουμε να έχουμε ένα σοσιαλιστή επιπλέον. Νομίζω ότι είναι εύκολο να το αποφύγουμε να ψηφίσει ένα λιγότερο. Δεν βλέπει το Προεδρείο ποιο ψηφίζει και ποιο δεν ψηφίζει. Απλώ το Προεδρείο βλέπει ότι υπάρχει μια ψήφο παραπάνω. Εκτό μικροφώνου το σχόλιο τη κυρία Γκαρσία. Εσείς είσαστε υπεύθυνοι για την ψηφορία σε σχέση με το ποιοι μπορούν και ποιοι δεν μπορούν να ψηφίσουν. Και να σας πω την αλήθεια δεν μπορώ να σας απαντήσω γιατί δεν άκουσα τι λέτε. Λοιπόν, 82 για νιωστή φορά. Vamos a intentar mantenerlo así durante la votación. Λοιπόν, άρχεται η ψηφορία για την 82. Ρετσαθάδα. Απορρίπτεται. Τροπολογία 83. Άρχεται ψηφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 86. Άρχεται η ψηφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Περνάμε στην 88. Αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 89. Άρχεται η ψηφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 91. Άρχεται η ψηφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 92. Συγγνώμη, 90, 90. Ψηφίζεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 92. Πέρας. Απορρίπτεται. MV8. Ψηφίζεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Έχει αποσυρθεί η 94 της κυρίας Μπιλμπάου. Περνάμε στην 95. Άρχεται η ψηφορία. 95. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβασμός 1. Άρχεται η ψηφορία. Πάλι έχουμε έναν σοσιαλιστή πλέον. Για να δούμε. Δεν ξέρω πώς είναι δυνατόν να μην υπάρχουν πλέον τροποποίησεις. Εντάξει, αυτό λέει εδώ το μηχάνημα, ότι υπάρχει ένας παραπάνω. Κυρία Μιλάνα, δεν θα κάτσω τώρα να τσακωθώ μαζί σας. Είναι ηλεκτρονική η ψηφοφορία, όσο και εσείς αν θέλετε εδώ τώρα να το αμφισβητήσετε. Μπορούμε να κάνουμε κάτι έτσι ώστε να μην υπάρχουν ε, τροποποιήσεις. Να επαναλάβουμε. Συμβιβασμό ένα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Αγκρίνεται. Να περάσουμε στο συμβασμό 2. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβασμό 3. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβασμός 3α. Αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 108. Άρχεται η ψηφορία. Thank ε, down. Non, euh, Claude, oui, 108. Après les 13 bis, 108. On n'est pas trop vite. ¿Cuál es el problema? Después de los compromisos. Ποιο είναι το πρόβλημα. Μετά την NV11, βλέπετε, είναι η τροπολογία 108. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Απορρίπτεται. 111. Άρχεται ψηφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβασμός 4. Αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβασμός 5. Άρχεται ψηφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 115 τροπολογία. Αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. 121. Αρχίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβασμό 6. Άρχεται η ψηφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 130. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 132. Άρχεται ψηφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 135. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 133. Άρχεται η ψηφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβασμός 7 με τμήματική ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα. Αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Αρχίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Περνάμε στην 141. Αρχή. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβασμός 7α. Άρχεται η ψηφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 142. Άρχεται η ψηφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 145. Άρχεται η ψηφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 147. Πέρας. Απορρίπτεται. 148. Αρχή. Πέρας. Απορρίπτεται. 151. Αρχή. Πέρας. Απορρίπτεται. 12-12. 149. Αρχή. Πέρας. Απορρίπτεται. 150. Άρχεται η ψηφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 152. Αρχή. Πέρας. Απορρίπτεται. 17 Αρχή. Τέλος. Απορρίπτεται. 153. Άρχεται η ψηφορία. αέρας Απορρίπτεται. 154. Πέρας. Απορρίπτεται. 13. Πέρας. Εγκρίνεται. 159. Συγγνώμη. 162 λέει ο πρόεδρο. Πάμε στην 162. Αρχή. Πέρα. Αγκρίνεται. Συμβασμός 8. Αρχή. Πέρα. Αγκρίνεται. 168. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας.

Εγκρίνεται. 176. Αρχή. Πέρας. Απορρίπτεται. 177. Αρχή. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβασμός 9 σε δύο μέρη. Πρώτο τμήμα. Αρχή. Πέρας. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. Ας περάσουμε στην 187. Στην τροπολογία 187 αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. 188. Αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. 190. Άρχεται ψηφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 192. Αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. 15. Συγγνώμη, συμβιβασμός παριθμών 10. Αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 15. Αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 199. Αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. 201. Αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. 202. Πέρας. Εγκρίνεται. 204. Πέρας. Εγκρίνεται. 205. Πέρας. Απορρίπτεται. NV22. Και. Πέρας. Απορρίπτεται. 206. Πέρας. Δεν κρίνεται. 207. Πέρας. τα κρίνεται. 208. Πέρας. Εγκρίνεται. 29. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβασμός 11. Απροβάρα. 200. Εγκρίνεται. 214. Πέρας. Εγκρίνεται. 215. Πέρας. Εγκρίνεται. Πασαμος 23 Περνάμε στην MB23. Πέρας. Απορρίπτει. 219. Πέρας. Εγκρίνεται. 220. Πέρας. Εγκρίνεται. 221. Πέρας. Εγκρίνεται. 2022. Πέρας. Γκριντ. 223. Πέρας. Απορρίπτεται. 224. Πέρας. Γκρίνεται. Συνδεσμος 12. Πέρας. Γκρίνεται. 226. Πέρας. Εγκρίνεται. 232. Πέρας. Απορρίπτεται. 234. Πέρας. Απορρίπτεται. 2.35. Πέρας. Απορρίπτεται. 238. Πέρας. Απορρίπτεται. 2.37. Πέρας. Απορρίπτεται. 239. Πέρας. Απορρίπτεται. 241. Πέρας. Γκρίνεται. 16. Πέρας. Γκρίνεται. 243. 244 διορθώνει ο πρόεδρος. 244. Πέρας. Εγκρίνεται. 245. Πέρας. Εγκρίνεται. 246. Πέρας. Εγκρίνεται. 247. Πέρας. γκρίνεται 248. Πέρας. γκρίνεται 249. Πέρας. γκρίνεται 250. Πέρας. γκρίνεται Κύριος Καντέκ, προφορική τροπολογία. Δεν χρειάζεται να μας τα εξηγήσετε. Την έχετε όλοι. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Γκρίνεται. 251. Πέρας. Εγκρίνεται. 252. Πέρας. Εγκρίνεται. 253. Πέρας. Εγκρίνεται. 254. Πέρας. Απορρίπτεται. 125. Πέρας. Απορρίπτεται. 255. Πέρας. Εγκρίνεται. 257. Πέρας. Εγκρίνεται. 258. Πέρας. Απορρίπτεται. 260. Πέρας. Εγκρίνεται. 261. Πέρας. Απορρίπτεται. 262. Πέρας. Εγκρίνεται. 263. Πέρας. Εγκρίνεται. 264. Πέρας. Εγκρίνεται. 265. Πέρας. Εγκρίνεται. 266. Πέρας. Εγκρίνεται. 267. Πέρας. Εγκρίνεται. 268. Πέρας. Εγκρίνεται. 269. Ρετσαθάδα. Απορρίπτεται. 270. Πέρας. Απορρίπτεται. Ένβη. 28. Πέρας. Εγκρίνεται. 271. Πέρας. Απορρίπτεται. 272. Πέρας. Απορρίπτεται. Ένβη 29. Πέρας. Εγκρίνεται. 274. Πέρας. Εγκρίνεται. 278. Συγγνώμη. Πάμε στην 277. Πέρας. Rechazada. 279. Comienza. 279. Αρχή. Πέρας απορρίψετε. 282. Σιέρα. Πέρας. Εγκρίνεται. Πασάμος αλλά 285. 285. 285. Αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. 286. όχι. 287. Πέρας. Απορρίπτεται. MP30. Αρχή. Πέρας. Απορρίπτεται. 288 αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. 289 αρχή. Πέρας. Απορρίπτεται. 2,90. Αρχή, πέρας. Εγκρίνεται. 2,93. Αρχή. Πέρας. Απορρίπτεται. 19. Αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. 2,94. Πέρας. Green. 2. 299. Αρχή. Πέρας. Απορρίπτεται. 300. Αρχή. Πέρας. Απορρίπτεται. 301. Αρχή. Πέρας. Απορρίπτεται. 302. Αρχή. Πέρας. Απορρίπτεται. 303. Αρχή. Πέρας. Απορρίπτεται. 304. Αρχή. Πέρας. Απορρίπτεται. Συγγνώμη, κυρία Λοβάν. You're going too fast. Πάτε πάρα πολύ γρήγορα. Συγγνώμη. A ver, nos hemos quedado 300... 304. Να επαναλάβουμε την ψηφοφορία για την 304 τροπολογία. Αρχή. Πέρας. Απορρίπτεται. 305. Αρχή. Πέρας. Απορρίπτεται. 20. Αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. 306. Αρχή. Πέρας. Απορρίπτεται. Εμμήντα 308. 308. Αρχή. Πέρας. Απορρίπτεται. 21. Αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. 309. Αρχή. Πέρας. Απορρίπτεται. 310. Αρχή. Τερμίνα. Πέρας. Απορρίπτεται. 3.11. Αρχή, πέρας. Απορρίπτεται. 312. Αρχή. Πέρας. Απορρίπτεται. 313. Αρχή. Πέρας. αγκρίνεται. 314 αρχή. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβασμός 13. Σε δύο μέρη. Πρώτο τμήμα. Αρχή. Πέρας. αγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Αρχή. Πέρας. Απορρίπτεται. Περνάμε στην 317. Αρχή. Πέρας. Απορρίπτεται. 318. Αρχή. Πέρας. Απορρίπτεται. 319. Αρχή. Πέρας. Απορρίπτεται. 320. Αρχή. Πέρας. Απορρίπτεται. 321. Αρχή. Πέρας. Απορρίπτεται. NV33. Αρχή. Πέρας. Απορρίπτεται. 322. Αρχή. Πέρας. Απορρίπτεται. Λοιπόν, από κοινού 323 και 325. Αρχή. Πέρας. Απορρίπτονται. 324. Αρχή. Πέρας. Απορρίπτονται. 326 αρχή. Πέρας. Απορρίπτεται. 327 αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. 330 αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. 331. Συγγνώμη. 334. Αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. 335. Αρχή. Πέρας. Απορρίπτεται. 336. Αρχή. Πέρας. Απορρίπτεται. 337 αρχή. Πέρας. γκριντ. 338 αρχή. Πέρας. γκριντ. 340 αρχή. Πέρας. Απορρίπτεται. 341 αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. 342. Αρχή. Πέρας. Απορρίπτεται. 347. Αρχή. Πέρας. Απορρίπτεται. 344. Αρχή. Πέρας. Απορρίπτεται. 345 αρχή. Πέρας. Απορρίπτεται. 346 αρχή. Πέρας. Απορρίπτεται. MP34 αρχή. Πέρας. Απορρίπτεται. MP35 αρχή. Πέρας. Απορρίπτεται. 348. Αρχή. Πέρας. Απορρίπτεται. 349. Αρχή. Πέρας. Απορρίπτεται. 350. Πέρας. Εγκρίνεται. 351. Αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβασμός 14. Αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 360. Αρχή. 360. Αρχή. Αέρας. Απορρίπτεται. 361. Αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. 362. Πέρας. Απορρίπτεται. 363. Πέρας. Απορρίπτεται. 364. Αρχή. Πέρας. Απορρίπτεται. 365. Αρχή. Πέρας. Απορρίπτεται. 366 αρχή. Ένας. Εγκρίνεται. 38 αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. 367 αρχή. Πέρας. Απορρίπτεται. 368 αρχή. Πέρας. Απορρίπτεται. 369. Αρχή. Πέρας. Απορρίπτεται. 370. Αρχή. Πέρας. Απορρίπτεται. 371. Πέρας. Απορρίπτεται. 372. Αρχή. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβασμός 15 σε δύο μέρη. Πρώτο τμήμα, έρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Περνάμε στην 300. 77. Άρχεται η ψηφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Λοιπόν, προφορική τροπολογία για το 41 παραγωγός 1, σημείο ΔΕΛΤΑ άλφα, νέο, άρχεται η ψηφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 16, Αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβασμός 17. Αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. 1.39. 386 λέει τώρα ο πρόεδρος. Άρχεται η ψηφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Tres nueve, nueve. Περνάμε στην 399. 399. En, comienza. Αρχή. Cierra. Πέρας. Aprobada. Εγκρίνεται. 27. Αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται.

αρχή, πέρας, εγκρίνεται. 414, αρχή, πέρας, εγκρίνεται. 416, αρχή, πέρας, εγκρίνεται. 417, αρχή, Έρας. Εγκρίνεται. 419. Αρχή. Έρας. Εγκρίνεται. 420. Αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. 422. Αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. 423. Αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. 424. Αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. 425. Αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. 426. Αρχή. Πέρας. Απορρίπτεται. 427, Αμπρε. 427. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 30. Αρχή, πέρας. Απορρίπτεται. 430 αρχή, πέρας. Εγκρίνεται. 431 αρχή, πέρας. αγκρίνεται. 443. 33, με συγχωρείτε. Πέρας. αγκρίνεται. 434, αρχή. Πέρας. Απορρίπτεται. 435 αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 31. Μετά την 46. 31. Αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. 43. Πέρας. Εγκρίνεται. 445. Αρχή. Πέρας. Απορρίπτεται. 446. Αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. 447. Πέρας. Εγκρίνεται. 448. Αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. 449, 350, 351 σε μπλοκ. Αρχή. Πέρας. Απορρίπτονται. 454. Αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. 455 αρχή. Πέρας. Απορρίπτεται. 32. Αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. 457. Αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. 460. Αρχή. 460. Πέρας. Εγκρίνεται. Πάμε στα παραρτήματα. 461. Αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. 462. Αρχή. Πέρας. Απορρίπτεται. 463. Αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. 464. Αρχή πέρας, εγκρίνεται. 465 αρχή. 466. 466 λέει ο πρόεδρος. Πέρας. Εγκρίνεται. Λοιπόν, καταπίπτει 467, περνάμε στα εκτιμώντας. 34, αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. NV1. Αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. Ένα. Αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. 35. Αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. 36. Αρχή. Αέρας. Εγκρίνεται. 37. Αρχή. Αέρας. Εγκρίνεται. 38. Αρχή. Αέρας. Απορρίπτει. 39. Αρχή. Ένας Εγκρίνεται. Συμβασμός 19. Αρχή. Ένας Εγκρίνεται. Περνάμε στην ένβη 3. Αρχή. Ένβη 3. Υπάρχουν τρία τροπολογία. Αρχή, πέρας. Απορρίπτεται. Τέσσερα. Αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. 46. Αρχή. Πέρας. Απορρίπτεται. 47. Αρχή. Πέρας. Απορρίπτεται. 48, αρχή. Πέρας. Απορρίπτεται. NV3, αρχή. Πέρας. Απορρίπτεται. 49, αρχή. Πέρας. Απορρίπτεται. 50. Πέρας. Απορρίπτεται. NV4. Αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. 51. Αρχή. Τέλος. Απορρίπτεται. 52. Αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. 189 αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. 53 αρχή. Πέρας. Απορρίπτεται. 54 αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβασμός 20 αρχή. Αποχές. Εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 57. Αρχή. Πέρας. Απορρίπτεται. 58. Αρχή. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 6. Αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 7. Αρχή. Πέρας. Τροπολογία 7. Εγκρίνεται. Τροπολογία 8. Αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. 61. Αρχή. Πέρας. Απορρίπτεται. 65. Συγγνώμη. 62. 62. Αρχή. Πέρας. Απορρίπτεται. 66. Αρχή. Πέρας. Απορρίπτεται. 63. Αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. 67. Αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. 68. Αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. 69. Αρχή. Αέρας. Απορρίπτεται. 70. Αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. 71. Αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. Να περάσουμε τώρα στο να ψηφίσουμε την νομοθετική πρόταση έτσι όπως τροποποιήθηκε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Και τέλος, να ψηφίσουμε το ψήφισμα, την πρόταση ψηφίσματος. Αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται με ευρύτατη πλειοψηφία. 24 προς 1. Ολοκληρώσαμε λοιπόν. Συγχαρητήρια και στον κύριο Στίβενσον. Και καθώς κινηθήκαμε γρήγορα, θέλετε να κάνουμε ένα διάλειμμα 5 λεπτών. 5-7 λεπτά. Bueno. que vamos tomando asiento. We start. Θα συνεχίσουμε παρακαλώ. Sin prisa, pero sin pausa. Θα σπεύσουμε βραδέως για να τα κάνουμε όλα σωστά. Bien, pasamos a la votación. Si ya estamos todos, yo creo que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 Είπαμε να σταματήσουμε για 5 λεπτά, είναι 10, σημείο 5 για τον κανονισμό σχετικά με την ε, διατήρηση των αλλιευτικών πόρων στα πλαίσια της κοινή αλλιευτικής πολιτικής, ε, έκθεση του κυρίου Χάγκλουντ. Αν δεν έχετε ερωτήσεις ε, πριν από την ψηφοφορία και συμφωνείτε, ας αρχίσουμε ευθύ αμέσως. Την προηγούμενη, την προηγούμενη την καταφέραμε. Θα προσπαθήσουμε τώρα να είμαστε εξίσου καλοί τουλάχιστον. Ε, Αρχίζουμε. Η τροπολογία 13. Όχι, διορθώνει ο Πρόεδρος. 12. Ωραία, αρχίζουμε πάλι. 12. Τροπολογία 12 αρχή, πέρας, εγκρίνεται. 17. Όχι, αφού έχει εγκριθεί 12, δεν θα ψηφίσουμε τη 17. Μην 14. 14. Τροπολογία 14, αρχή. σε δύο μέρη. Με συγχωρείτε. Πρώτο μέρος. Πέρας. Απορρίπτεται το πρώτο τμήμα. Δεύτερο τμήμα. Αρχή. Πέρας. Αγκρίνεται το δεύτερο τμήμα. Τροπολογία 11. Αρχή. Τέλος. Δεν κρίνεται. 13. Αρχή. Πέρας. Δεν κρίνεται. Τροπολογία 15. Αρχή. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβασμός 11. Αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 19. Αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 21. Αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 22. Αρχή. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 20. Αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 24. Αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. 25, αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. 26, αρχή. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβεσμός 1, αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. Πάμε στο 27. Σε δύο μέρη τροπολογία 27. Πρώτο τμήμα. Αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Αρχή. Πέρας. απορρίπτεται. Τριάντα πέντε. Τροπολογία τριάντα πέντε. Αρχή. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 36, αρχή. Πέρας. Απορρίπτεται. 37, αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβασμός 2. Αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 43 σε δύο μέρη. Πρώτο τμήμα, αρχή. Συγγνώμη, δεύτερο τμήμα λέει ο πρόεδρος τώρα. Το δεύτερο τμήμα, γιατί καταπίπτει το πρώτο. 43 δεύτερο τμήμα λοιπόν, αρχή. Πέρας. Απορρίπτεται. Σαράντα τέσσερα. Αρχή. Πέρας. Λοιπόν, ψηφίσαμε το δεύτερο τμήμα της 43. Ah, it's 44. 44. Ah, okay. Ah, ah, okay. That's it. 44. 44. Αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. 45. Αρχή. Πέρας. Απορρίπτεται. 46. Αρχή. Πέρας. Απορρίπτεται. 47. Αρχή. Πέρας. Απορρίπτεται. Πενήντα ένα. Αρχή. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβασμός τρία. Αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. Σαράντα εννέα. Αρχή. Πέρας. Απορρίπτεται. 53. Αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. Να ψηφίσουμε τώρα σε μπλοκ τις ε, τροπολογίες 54 και 56. Αρχή. Πέρας. Απορρίπτεται. 55. Αρχή. Πέρας. Απορρίπτεται. σε μπλοκ την 57 και την 58. Αρχή. Πέρας. Απορρίπτεται. Περνάμε στο συμβιβασμό υπαριθμών 4 με τη μαματική ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα αρχή, πέρας. Πέρας, εγκρίνεται. Να περάσουμε. Σε μπλοκ ψηφίζουμε τις τροπολογίες 65-73, αρχή, Yeah. It's in block 65. Σε μπλοκ 65-71-73. Εντάξει. Αν, προσ... αν προτιμάτε να τα λέω και στα αγγλικά. Σε μπλοκ 65-71-73. Εντάξει. Πέρας. Απορρίπτεται. 66. Υπάρχει. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβασμός 8. Ξεχωριστή ψηφορία, κομματική ψηφορία, πρώτο τμήμα, αρχή, πέρας. Εγκρίνεται, δεύτερο τμήμα. Αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. Now we go to 67. Yes. Yes. 67. 67. Ξεκινάμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 70. Αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβασμός 5. Αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. Εβδομήντα έξι. Αρχή. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβασμός έξι. Αρχή. Αέρας. Εγκρίνεται. Τεχνολογία 80. Αρχή. Αέρας. Απορρίπτεται. Συμβασμός 7. Αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 86, αρχή. Πέρας. Απορρίπτεται. 87, αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. 88. Αρχή. Πέρας. Απορρίπτεται. 89. Αρχή. Πέρας. Απορρίπτεται. 91. Αρχή. Αέρας απορρίπτεται. 94, αρχή. Πέρας. Απορρίπτεται. 92. Αρχή. Πέρας. Απορρίπτεται. 93. Αρχή. Πέρας. Απορρίπτεται σε μπλοκ 95, 96, 97. Αρχή. Πέρας. Απορρίπτεται. 98. Αρχή. Πέρας. Απορρίπτεται. 99. Αρχή. Αέρας. Απορρίπτεται. Εκατό. Αρχή. Πέρας. Απορρίπτεται. 101. Αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. 102. Αρχή. πέρας απορρίπτεται 103 αρχή πέρας εγκρίνεται 104 αρχή πέρας εγκρίνεται 105 αρχή πέρας απορρίπτεται 106 αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. 107 αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. 108 αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. Εκτιμώντας ένα Αρχή. Εγκρίνεται. Δύο. Πνευματική ψηφορία, πρώτο τμήμα. Αρχή. Πέρας, απορρίπτεται. Τμήμα δύο. Αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. Εκτιμώντας γάμα, τροπολογία 3. Ποιοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 4. Ποιοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβασμός 9. Αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. 6. Τιμώντας 6. Τιμώντας ε, τροπολογία 6. Τροπολογία 6, αρχή, πέρας, απορρίπτεται. Τροπολογία 7, αρχή, πέρας, εγκρίνεται. Συμβασμός 10. Αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 9. Αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. Και τέλος να ψηφίσουμε υπέρ της πρότασης ψηφίσματος που τροποποιήθηκε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία. Συγχαρητήρια κύριε Χάγκα. Και αφού ολοκληρώσαμε και αυτό το σημείο, συγχαρητήρια. Να περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημερικής διάταξη. ψηφοφορία για τα Ευρωπαϊκά Ταμεία και κατάργηση του κανονισμού 1083 του 2006. Ο κύριος Μπεσέτη είναι ο εισηγητής. Να συνεχίσουμε λοιπόν. Τροπολογία 1. Ah. Ψήσατε. Πέρας. Εγκρίνεται. Δύο. Αρχή. Ψήσατε. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 16. Αρχή. Ψηφίσατε. Εγκρίνεται. Τροπολογία 17. Αρχή. Αγκρίνεται. Τροπολογία 3. Αρχή. Ε, πέρας. εγκρίνεται. Τροπολογία 4, αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 18, αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5, αρχή. Εγκρίνεται. Τροπολογία 6. Αρχή. Πέρα. Εγκρίνεται. Τροπολογία 19. Αρχή. Πέρα. Εγκρίνεται. 20. Αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. 7. Αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. 21. Αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. 8. Αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. 9. Αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. Δέκα. Αρχή. Αέρας. Εγκρίνεται. Έντεκα. Αρχή. Αέρας. Απορρίπτεται. Δώδεκα. Πέρας. Εγκρίνεται. 22. Αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. 23. Αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. 24. Αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεκατρία. Αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεκατέσσερα. Αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεκαπέντε. Αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τη γνωμοδότηση στο σύνολό τη. Αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. Ευχαριστούμε πολύ. Συγχαρητήρια κύριε Μπεσέτ. Στη συνέχεια η ειδική 12.2011. συντάκτη είναι ο κ. Μιλάνα. Να συνεχίσουμε. Τροπολογία 1. Αρχή. Πέρας. Απορρίπτεται. Δύο. Αρχή. Πέρας. Απορρίπτεται. Σε μπλοκ 3, 4, 5 και 6. Αρχή. Πέρας. Εγκρίνονται. Συμβαστική τροπολογία 1. Ε, αρχή. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 7. Αρχή. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 10. Αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 9. Αρχή. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 11. Αρχή. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 12. Αρχή. Πέρας. Απορρίπτεται. 13. Πέρας. Απορρίπτεται. 14. Αρχή. Τέλος. Εγκρίνεται. Σε μπλοκ. Τροπολογίες 15 και 16. Αρχή. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 17. Αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. Σε μπλοκ 18, 19 και 20 αρχή. Να τις αρχίσουμε. 18, 19, 20. Πέρας. 22. Τμηματική ψηφοφορία, πρώτο τμήμα, αρχή. Ξαναρχίζουμε. Χωρίς τη ψηφοφορία, τροπολογία 22, πρώτο τμήμα. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Αρχή. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 23. Αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. 24. Πέρας. Απορρίπτεται. 25. Πέρας. Απορρίπτεται. 27. Πέρας. Απορρίπτεται. 27. ψηφίσαμε την 27, ήταν 26. Να επαναλάβουμε, 26. Συγγνώμη. 26. Πέρας. Εγκρίνεται. 27. Αρχή. Πέρας. Απορρίπτεται. 28. Αρχή. Πέρας. Αγκρίνεται Συμβασμός 3. Αρχή. Πέρας. Αγκρίνεται Απολογία 30. Αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. 31. Πέρας. Εγκρίνεται. 33. Πέρας. Απορρίπτεται. 34. Πέρας. Εγκρίνεται. 32. Αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται σε μπλοκ 36 και 37. Αρχή. Πέρας. Απορρίπτεται. 38. 14, ne? Right? 40. 40. Amendment 40. 40, λέει ο πρόεδρος. Πέρας. Υιοθετείτε. 41. Πέρας. Απορρίπτεται. 42. Πέρας. Εγκρίνεται. 43. Συγγνώμη, 44. 44. Πέρας. Εγκρίνεται. 46. Πέρας. Εγκρίνεται. 47. Πέρας. Εγκρίνεται. 48. Πέρας. Απορρίπτεται. 49. Πέρας. Γκρίνεται. 50. Πέρας. Γκρίνεται. 51. Πέρας. Απορρίπτω. 52. Πέρας. 53. κρίνεται 52, 53. Πέρας. Απορρίπτεται 54. Αρχή. Πέρας γκρίνεται. 55. Π.χ. Πέρας. γκρίνεται. 56. Αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. 57. Αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. 58. Αρχή. Πέρας. Απορρίπτεται. 59. Αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα το σύνολο της πρότασης κειμένου. Άρχεται η ψηφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια. Κύριε Μπεσέτλη, ο πρόεδρος. Κύριε Μιλάνα, διορθώνει. Bueno, hemos terminado. Ολοκληρώσαμε την ψηφοφορία. Σας ευχαριστώ όλους. Ευχαριστώ όλους τους βουλευτές. Πολύ πιο γρήγορα από ό,τι είχαμε προβλέψει. Έτσι λοιπόν έχετε περισσότερο χρόνο για το διάλειμμα και στις 3 ακριβώς ε, θα ξαναρχίσουμε να είστε ακριβείς παρακαλώ, θα τα ξαναπούμε στην ίδια αίθουσα, γιατί έχουμε τη μήνυα ακρόαση. Και κατόπιν ε, θα έρθει και η κυρία Επίτροπος και θα δούμε και τα υπόλοιπα σημεία στην ημερήσια διάταξη. Σας ευχαριστώ, τα ξαναλέμε στις 3 ακριβώς. Gabriel. Thank you. good.